Αγαπητοί συνάδελφοι, σα ζητώ συγγνώμη για αυτήν την καθυστέρηση. Σε κάθε περίπτωση, με ιδιαίτερη χαρά, ξεκινάμε αυτό το απόγευμα με την δημόσια ακροασή μα ε, όσον αφορά το ρόλο των δημόσιων συγκοινωνιών σε αεροκατοικημένε περιοχές και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε μαζί μα τέσσερι εμπειρογνώμονε. Σα καλωσορίζω στην Επιτροπή μα. Η κινητικότητα, το γνωρίζετε, αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα για την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και αποτελεί έναν ουσιαστικό λόγο για τον οποίο δική μας η Επιτροπή αποφάσισε να διοργανώσει τη δημόσια κρόαση με το θέμα αυτό και πραγματικά θα έλεγα ότι είναι το σημαντικότερο καύσιμο της ε, οικονομικής ανάπτυξη, η κινητικότητα αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να προωθήσουμε την κινητικότητα παντού έχοντας κατά νου και την κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά καταλήγουμε στο αντίθετο της κινητικότητα στην ακινησία. Που ακινησία σημαίνει ότι δεν βγαίνει κανείς έξω, δεν βλέπει τον κόσμο, δεν συμμετέχει στα κοινά, δεν συμμετέχει στην κοινωνική οικονομική ζωή. Πέρα από την κοινωνική αυτή αδικία. Έχουμε και την κλιματική αλλαγή που μας επιβάλλει να δημιουργήσουμε αποτελεσματικά μέσα δημοσίων μεταφορών, αν πραγματικά θέλουμε να βρούμε μια εναλλακτική λύση στην αποκλειστική χρήση των ε, αυτοκινήτων. Όπως ξέρετε, χρησιμοποιούνται πάρα πολύ, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο και πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλά νοικοκυριά εξαρτώνται από το αυτοκίνητο, που σύν τις άλλες είναι και ένα δαπανηρό μέσο μεταφοράς. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε μέσω της ακρόασης αυτής να φωτίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν θετήσει διάφορες χώρες, προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες στις πιο απομακρυσμένες και αεροκατοικημένες περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να σας παρουσιάσω την κυρία Πάουλα Τέλες. Είστε πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Κινητικότητα στις πόλεις και στα χωριά, Ινστιτούτου της Πορτογαλίας. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να καλωσορίσω επίσης τον κύριο Ματίας Λάνταν, ο οποίος είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των δημοσίων συγκοινωνιών και μεταφορών στην περιοχή Βάρλαν της Σουηδίας. Καλώς ήλθατε επίσης στην Επιτροπή μας. Να καλωσορίσω επίσης τον κύριο Ρωμάν Στερμπάι Πίκουρο, καθηγητή στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Τσεχίας, υπεύθυνο επίσης για την ανάπτυξη των ε, τσεχικών δημοσίων σιδηροδρομικών υποδομών και να καλωσορίσω επίσης και τον κύριο Κρέστιανσεν, ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής της βελγικής Mobile Mobiel21. Αγαπητοί εμπειρογνώμονες, αγαπητοί μας καλεσμένοι, έχετε 10 λεπτά έκαστο στη διάθεσή του, προκειμένου να μας παρουσιάσετε με τρόπο περιληπτικό, συνθετικό, τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στις χώρες σας και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η συζήτηση με τους συναδέλφους. Ξεκινάμε με τις κυρίες, γιατί έτσι ήθιστε. Κυρία Πάουλα Τέλες, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ για να εκπροσωπήσω τη χώρα μου και ε, το Ινστιτούτο μας είναι ιδιωτικό Ινστιτούτο. Έχουμε εργαστεί με την κυβέρνηση της Πορτογαλίας ε, για πάνω από 15 χρόνια και με τους Δήμους ε, της Πορτογαλίας ε, προωθώντας τις πολιτικές βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η κινητικότητα σήμερα θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα έλεγα ότι το, θέμα της στέγασης που είναι μία από τις πρώτες πολιτικές είναι στις ανησυχίες μας θα έλεγα ότι και η κινητικότητα ε, στις ε, διάφορες ε, επικράτειες είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα μάθω πολλά, θα μάθετε πολλά από αυτά που θα πω, γιατί είμαστε πολύ μικρή χώρα, αλλά θα ξεκινήσω τώρα την παρουσίασή μου. Η χώρα μας είναι πολύ μικρή, όπως σας είπα είναι στην περιφέρεια της ε, Ευρώπης, βρισκόμαστε στην Βυρική Χερσόνησο δίπλα από την Ισπανία. Όμως, ε, παρόλο που είναι μικρή η χώρα, είναι πολύ διαφοροποιημένη σε σχέση με τις διάφορες περιφέρειες. Έχει πολύ μεγάλες διαφορές από το βορρά στο νότο σε ό,τι αφορά ε, και τον αριθμό των διοικητικών μονάδων Έχουμε 10 εκατομμύρια κατοίκου και τα 3 τέταρτα του πληθυσμού μα ε, ζουν ε, σε παραθαλάσσιε περιοχέ. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα λοιπόν στο εσωτερικό που είναι κοντά στην Ισπανία όπω βλέπετε εδώ. Το 22% του πληθυσμού σήμερα είναι πάνω από 65 ετών. Έχουμε δηλαδή ένα πληθυσμό ιδιαίτερα γερασμένο. Το 11% είναι άνω των 75 ετών. Το 17% έχει τουλάχιστον ε, μια σωματική αναπηρία. Πρόκειται λοιπόν για μια χώρα πρέπει να εργαστεί πολύ γρήγορα για να μπορέσει να φτάσει την ταχύτητα που θέλει και ε, πρέπει να εργαστούμε σε δύο ταχύτητες όπως θα πούμε και εδώ σήμερα η Πορτογαλία ε, δεν ε, ε, έχει ουσιαστικά μία παγκόσμια ταξινόμηση για την ε, έννοια των αεροκατοικημένων περιοχών. Ε, βλέπετε ότι είχαμε κάποιες ευρωπαϊκές πολιτικές του 2016. Εκπονήσαμε ένα εθνικό πρόγραμμα για την εθνική συνοχή. Βασιστήκαμε σε πολλά κριτήρια, την δημογραφία, την πυκνότητα του πληθυσμού, τις εγκαταστάσεις του πληθυσμού, τα, χαρακτηριστικά, τα φυσικά χαρακτηριστικά της επικράτειας, την τα κοινωνικομικά χαρακτηριστικά, την προσβασιμότητα όμω έχουμε διάφορα προβλήματα στις διάφορες περιφέρειες. Ε, Παραδείγματο χάρη έχουμε απώλεια του πληθυσμού και αύξηση του, της του πληθυσμού. Έχουμε πληθυσμό με λιγότερα προσόντα, όλο ένα και περισσότερο. Ε, επίσης ε, τα ευρωπαϊκά, συγγνώμη, αστικά κέντρα δεν έχουν τι επιθυμητές διαστάσει. Γενικά έχουμε ε, στις αεροκατοικημένες περιοχές, χαμηλή οικονομική δραστηριότητα, είναι όλο ένα και πιο ανενεργός ο πληθυσμός, καθώς γυράσκει και έχουμε μικρά δίκτυα συμπράξεων, αδύναμα δίκτυα συμπράξεων ε, και διάφορα ποσοστά ε, πληθυσμού, μάλλον διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής ε, του πληθυσμού. Ε, αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, το ότι ο πληθυσμός δεν συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει ουσιαστικά μία πτώση στην Πορτογαλία. Έχουμε ε, αραιοκατοικημένες ε, περιοχές ε, και δυστυχώς υπάρχει και οικονομική ύφεση σε αυτές τις περιοχές. Επίσης, έχουμε δύο είδη Πορτογαλίας σε ό,τι αφορά την κινητικότητα. Μία Πορτογαλία που συνδέεται πάρα πολύ με το δικό δίκτυο και έχουμε ένα ισχυρό δίκτυο που συνδέει τις διάφορες επικράτειες, όμως περισσότερο συνδέει το βορρά προς τον, Νότο και επίσης, και επίσης ε, έχουμε και σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο όμως ε, δυστυχώς δεν προωθήθηκε πολύ από τις πολιτικές τις τελευταίες δεκαετίες επομένω. Ε, είναι πολύ περιορισμένες οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες ούτε καν δεν έχουμε τρένα υψηλής ταχύτητας και ε, ουσιαστικά είχαμε βασιστεί στις δημόσιες ε, μεταφορές αλλά δεν δόθηκαν κίνητρα και κατά τη διάρκεια πολλών ε, δεκαετιών δυστυχώς εγκαταλείφθηκε και σήμερα οι δημόσιες πολιτικές στην Πορτογαλία όπως ξέρετε θέλουν να προωθήσουν τους σιδηροδρόμους και εγώ θέλω να δω με ενθουσιασμό τι θα γίνει σύντομα. Λοιπόν, εδώ ε, συνεχίσουν να χάνουν πληθυσμό οι αεροκατοικημένες περιοχές ε, και φυσικά βλέπουμε μείωση στη ζήτηση για τις ε, τακτικές υπηρεσίες ε, μεταφορών. Υπάρχει αυξημένη πίεση για την οικονομική βιωσιμότητα και υπάρχει μείωση της ποιότητας ε, των υπηρεσιών και ο βασικός εξοπλισμός πρέπει να εξορθολογίζεται, το λένε και περισσότερο και φυσικά είναι πολύ πιο λίγα και τα μέσα μεταφοράς. Τι μπορούμε να πούμε τώρα με το τι συμβαίνει στη χώρα μας εμείς. Ε, έχουμε ε, την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη μεταφέραμε μέσα σε τρία-τέσσερα χρόνια στο εσωτερικό μας σύστημα. Εμείς ε, δεν κάναμε καλή δουλειά κατά τη γνώμη μου, δυστυχώς, ε, και πέρασαν ε, αυτά τα δέκα χρόνια και αυτή τη στιγμή τώρα προσπαθούμε να προλάβουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη δουλειά σε νέες συνθήκες. Υπάρχει ουσιαστικά αποκέντρωση των αρχών σε ό,τι αφορά τις μεταφορές έχουμε ε, κάποιες ε, αστικές ε, κοινότητες που συνδέουν ε, τους δήμους. Επομένως, έχουμε 18 συνολικά που έχουν διοριστεί και προσπαθούμε να τρέξουμε ενάντια στο χρόνο για να εφαρμόσουμε το νομικό καθεστώς των δημόσιων μεταφορών. Και Φυσικά αυτό προσπαθούμε για να μην μείνει η χώρα από τη μια μέρα στην άλλη χωρί μεταφορέ. Όμω λείπει ο σχεδιασμό. Δεν υπήρξε σχεδιασμό των δικτύων ούτε τη ε, προσαρμογή. Ε, ε, γιατί αυξανόταν και ο κόσμο στι πόλει και επίση απέτυχε ο σχεδιασμό τη κινητικότητα. Ο κανονισμό αυτή υλοποιήθηκαν, οι αρχέ εργάζονται προ αυτή την κατεύθυνση και επομένω αυτό είναι ε, κάτι ε, πολύ σημαντικό στην περίπτωση της Πορτογαλίας αλλά και άλλων χωρών. Ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί αυτές τις διαδικασίες. Όλοι θα πρέπει να εργαζόμαστε ομαδικά. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα σχεδιασμό των δικτύων. Και για να κλείσω, να σας μιλήσω για το ποιε θεωρώ εγώ ότι είναι οι καλές πρακτικές που έχουμε σε αυτή τη στιγμή και θα πρέπει υποχρεωτικά να μα απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια. Το πρώτο μέτρο. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναπτύξουμε υποχρεωτικά ε, τα βιώσιμα σχέδια ε, μεταφορών. Πρόκειται για αυτά τα σχέδια ε, που υλοποιούνται στις περισσότερες πόλεις ε, της Ευρώπης. Ε, μάλιστα έχω συμμετέχει σε πολλές τέτοιες συνεδριάσεις για το θέμα αυτό. Η Πορτογαλία πρέπει να είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη που δεν έχει τέτοια σχέδια και δεν το έχουμε υποχρεωτικά. Εμείς ε, λοιπόν ε, ε, πρέπει να θετήσουμε αυτά τα μέτρα και πρέπει να εργαστούμε και σε επίπεδο μέσων μεταφοράς αλλά και σε επίπεδο κόμβων και να πρέπει να εργαστούμε και σε θέματα επιμελητίας στις πόλεις και δεν ε, μιλάμε μόνο εδώ ε, για, τους, για τις μεταφορές μόνο, είχαμε προβλήματα και με τις στάσεις, ε, με τους κόμβους. Εμείς στην Πορτογαλία εκπονήσαμε ένα έγγραφο, ένα πρόγραμμα σχεδιασμού κινητικότητας, το οποίο λεγόταν Σχέδιο Βιώσιμων Μεταφορών ε, και αυτό ήταν για να βρεθεί η χρηματοδότηση. Έγινε μέσα σε τρεις μήνες σε Excel ε, και τα μέτρα ε, δυστυχώς όμως δεν ήταν τα κατάλληλα. Το δεύτερο μέτρο είναι η προώθηση των μεταφορών ευέλικτων μεταφορών για τις αεροκατοικημένες περιοχές. Δεν βλέπουμε άλλη λύση. Δεν είναι βιώσιμο μια τόσο μεγάλη χώρα ε, χαροκατοικημένη να μην ε, έχει συχνές συνδέσεις. Επομένως, πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ και αυτό κάνουμε στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή. Εδώ και μήνες μιλάμε για το θέμα αυτό και θέλουμε να προβλέψουμε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, ε, γιατί και εμείς θα πρέπει να μάθουμε από σας και να μπορέσουμε πράγματι να εφαρμόσουμε αυτές τις ευέλικτες μεταφορές. Τρίτο μέτρο, η σημασία της ε, προσβασιμότητας και του καθολικού σχεδιασμού. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε η Ευρώπη να μας βοηθήσει. Έχουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια, όμως ε, ε, εμείς θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στις επικράτειες όπου υπάρχει πραγματική γύρανση του πληθυσμού έχουμε τη μεγάλη υποδομή που είναι η πόλη. Θα πρέπει όλα αυτά να τα εντάξουμε σε ένα καθολικό σχεδιασμό και είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και από εδώ, γιατί δεν εργαζόμαστε μόνο στην Πορτογαλία, αλλά και από εδώ να ε, προσπαθήσουμε να εργαστούμε σε αυτό το τομέα. Το επόμενο μέτρο να προωθήσουμε ε, την ε, κατάσταση των υπηρεσιών, δεν έχουμε τους επαρκείς πόρους στις αεροκατοικημένες περιοχές. Και μάλιστα ε, μιλάμε και για την ιδιωτική οικονομία. Ε, πρέπει να συνεργαστούμε με τους ιδιώτες, να ιδρύσουμε υπηρεσίες που να είναι πιο ευέλικτες και ε, να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις αεροκατοικημένες περιοχές. Και πιστεύω εδώ σε επίπεδο υγείας, ε, παιδείας, ε, όπως και τις θεσμικές υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται αυτά. Τελευταίο μέτρο, πολύ σημαντικό στην Πορτογαλία, γιατί καθώς είναι τόσο μικρή η χώρα, έχουμε ε, ουσιαστικά μια ροκατοικημένη περιοχή που ε, γυτνιάζει με την Ισπανία. Έχουμε πολλές πόλεις που είναι κοντά στη Σαλαμάνκα, στο Βίγο, ε, στο Έλβα κτλ. Αλλά υπάρχει το σύνορο με την Ισπανία και δεν μπορούμε όμως στις μεταφορές να έχουμε αυτά τα σύνορα. Θα πρέπει ο σχεδιασμός να βασιστεί ε, στην ε, έννοια ε, της διασυνοριακότητας, δηλαδή να έχουμε ευρωπεριοχές. Και ουσιαστικά να υπάρχει μια σχέση μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας. Αυτά είναι τα πέντρα μέτρα που ήθελα να καταθέσω εδώ για να τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Έχουμε κάποια, τα εκπονεί τώρα η σημερινή κυβέρνηση και πολύ καλά και ουσιαστικά προσπαθούμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των κλιματικών αλλαγών και της απαρθρακοποίησης. Πολύ χρόνο έχει χάσει η Πορτογαλία, όμως αυτή τη στιγμή σε επίπεδο κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης γίνονται πάρα πολλά. Ε, εμείς προσπαθούμε να βάλουμε τα δυνατά μας για να μπορέσουμε να προλάβουμε ε, το τρένο και να υιοθετήσουμε τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές που υπάρχουν στις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ όλους και με στη διάθεσή σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή. Μας παρουσιάσετε πώς έχει κατάσταση στην Πορτογαλία. Τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Λαντά. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. thank you. Ευχαριστώ πολύ. Εργάζομαι για την αρχή δημοσίων μεταφορών στο Βέρμλαντ της Σουηδίας. Τώρα λειτουργεί. Ανάμεσα στη Στοκχόλμη και το Όσλο βρισκόμαστε στα δυτικά της Σουηδίας, ε, κοντά στα σύνορα με την Ορβηγία. Λίγα λόγια για το Δέρμπλαντ. Έχουμε περίπου 281.000 κατοίκους. 17,6 πληθυσμό ανά ε, τετραγωνικό χιλιόμετρο ε, με διακυμάνσεις από 62 ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο στο Κάλσταντ μέχρι 3 στο Τόσμπι. 50% ε, του πληθυσμού ζει μέσα στο Κάλσταρ και κοντά από αυτό, στα βόρεια ε, της λίμνης Βέρναν και το 40% ζει σε ε, περιοχές ε, αρεοκατοικημένες. Το 10% μένει σε χωριά με μέχρι χίλιους κατοίκους, ενώ το 30% μένει σε χωριά με λιγότερο από 200 κατοίκους. Αυτές είναι οι λευκές περιοχές του χάρτη. Αν κοιτάξουμε τις στάσεις λεωφορείων και σταθμούς τρένων, ε, καλύπτουμε περίπου το 90% του πληθυσμού. Ε, ζει δηλαδή σε απόσταση ε, το πολύ 1,5 χιλιόμετρο από στάση λεωφορείου ή σταθμό τρένου. Αλλά δεν εξυπηρετούνται πολυτακτικά όλες αυτές οι στάσεις και οι σταθμοί οι στάσεις ε, που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανεί για τις καθημερινές του μεταφορές ε, και μιλώ για μία αναχώρηση ανά ώρα ε, και στι δύο κατευθύνσεις, καλύπτουμε το 76 περίπου τα 100 του πληθυσμού. Εγώ θα σας μιλήσω λοιπόν για το υπόλοιπο 24%. Τι κάνουμε με αυτούς. κατασκευάζουμε ε, δημόσιες μεταφορές υψηλής χωρητικότητας ανάμεσα στις πόλεις και έχουμε κατόπιν ε, μέσα μεταφοράς χαμηλής χωρητικότητας ε, που μεταφέρουν τους κατοίκους σε, σε σημεία υψηλής μεταφοράς και επίσης κατασκευάζουμε και χώρους στάθμισης αυτοκινήτων σε αυτά τα κομβικά σημεία διότι όσοι έχουν τα πράγματα σήμερα, φαίνεται ότι αυτό είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για κάποιες περιοχές ε, να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες μεταφορές. Το μέλλον, το αύριο. Υπάρχει ανάγκη για συνεχή βελτίωση των δημοσίων μεταφορών ανάμεσα σε πόλεις. ώστε να έχουμε καλές μεταφορές ε, εντός ε, της ε, περιφέρειας αυτής και εξετάζουμε την λύση δημόσιες μεταφορές κατόπιν ζήτησης έξω από κάποιες βασικές αρτηρίες. Όλη η περιφέρεια έχει πρόσβαση σε δημόσιες μεταφορές που μπορεί να κλείσει κανείς εκ των προτέρων με το τηλέφωνό του ή με κάποια εφαρμογή στο έξυπνο κινητό του. Έτσι μπορεί να σας ε, μαζέψει κανείς από το σπίτι και να σας πάει στην πλησιέστερη πόλη. Εξετάζουμε επίσης τις δυνατότητες ε, για ε, μοίρασμα αυτοκινήτων σε κάποιες πιο αραιοκατοικημένες περιοχές, διότι έχουμε πολλές αρχές μεταφορών στην Σουηδία που επιτρέπουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Και αυτό γίνεται σε συνεργασία με άλλους φορείς και εταίρους. Σε δύο περιπτώσεις θα αναφερθώ. Η πρώτη περίπτωση είναι αυτή που λέγεται Traffic στα σουηδικά, ανοίγοντα τον δρόμο για το μέλλον. εξετάσαμε πόσο θα μας στοιχήσει να εκμεταλλευτούμε τη χωρητικότητα σε οχήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή για να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες. Και τα σχολικά λεωφορεία εξετάσαμε και τις υπηρεσίες ταξί. Εξετάσαμε τις περιπτώσεις αναπήρων ανθρώπων. Σε περίπτωση λοιπόν, ε, μάλλον τις ώρες που τα οχήματα αυτά δεν ε, χρησιμοποιούνται κανονικά, μήπως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλους σκοπούς και διαπιστώσαμε ότι πράγματι αυτό είναι δυνατόν και ότι θα στοιχήσει αυτό 800.000 το χρόνο για το σύνολο της περιφέρειας. Δεν είναι πολλά λεφτά αυτό. Αλλά βέβαια θα είναι κάπως περιορισμένες οι μεταφορές. Ε, θα πρέπει να κλείνει κανείς εκ των προτέρων ε, την ε, μεταφορά αυτή, πιθανότατα την προηγούμενη ημέρα και κάποιες ώρες της ημέρας δεν θα είναι διαθέσιμα τα οχήματα. Σε ένα χωριό το Φάγκερος θα εισάγουμε τώρα το καλοκαίρι ένα νέο σύστημα φαίνεται εδώ πέρα με το βέλος, έχει 442 κατοίκους και ε, πυκνότητα πληθυσμού 6,14 σαν τετραγωνικό χιλιόμετρο. Εξετάσαμε λοιπόν τις δυνατότητες συνδυασμένων μεταφορών ε, σε υπαίθριες περιοχές. Ε, πρόκειται για διαφορετική πλατφόρμα συνεργασίας ε, και παρέχει εναλλακτικέ λύσεις στην ιδιοκτησία αυτοκινήτου στις περιοχές αυτές. Και ενδιαφέρον εδώ είναι ότι συνομιλήσαμε πολύ με τους ε, κατοίκους του Φάγκερος, και εξετάσαμε τι ανάγκες καλύπτει ο στόλος των ΙΟΤΑΧΗ ε, σήμερα και πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες με δημόσιες μεταφορές. Πολύ ενδιαφέρουσα εδώ είναι η συνεργασία με ε, ένα τοπικό μπακάλικο. Εάν λοιπόν ε, μένει κανείς σε ε, χωριό που απέχει από το σούπερ μάρκετ μπορεί κανείς ε, να ε, κάνει την παραγγελία του και να σταλεί σε σε θηρίδες με ψήξη και να πάει κατόπιν να πάρει τα εμπορεύματά του από τις θηρίδες αυτές. Έτσι, δεν χρειάζεται να πάρει κανείς το αυτοκίνητό του μόνο και μόνο για να πάει να κάνει τα ψώνια του. Εξετάσαμε επίσης πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά τα σχολικά λεωφορεία. Σπανίως γνωρίζουμε σήμερα εάν κάθε πρωί θα, θα είναι γεμάτο το σχολικό, εάν κάθε παιδί θα πάει σχολείο. Διότι μπορεί το ένα παιδί να κοιμηθεί αλλού, μπορεί να αρρωστήσει. το οποίο σημαίνει ότι είναι δύσκολο να προσφέρουμε σε άλλους, σε, ε, σε άλλους κατοίκους σε τις ελεύθερες αυτές θέσεις. Ε, θέλαμε λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να ελέγχουμε καλύτερα εάν υπάρχει ε, διαθέσιμο δυναμικό, διαθέσιμος χώρος εντός των σχολικών λεωφορείων. Εδώ βλέπετε χάρτη που δείχνει τις διαδρομές των σχολικών λεωφορείων στο Φάγκερος. Ενώ τέλος ε, ε, αντιμετωπίζουμε και κάποιες προκλήσεις. Μία από τις μεγαλύτερες είναι φυσικά η χρηματοδότηση. Πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τις ε, καλές μαζικές μεταφορές σε αραιοκατοικημένες περιοχές, διότι είναι πολύ ακριβή η μεταφορά ανά άτομο. Θέλουμε λοιπόν νέα πιλωτικά προγράμματα για να δοκιμάσουμε νέες λύσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε το σύστημα. Πάντα μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Και όπως ανέφερα και πριν, ε, θα βλέπουμε μάλλον όλο και περισσότερους ε, ιδιωτικούς φορείς στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε ποια τμήματα της υπηρεσίας αυτής θα πρέπει να αποτελούν δική μας ευθύνη και τι θα πρέπει να κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να έχουμε ε, λειτουργικές και ποιοτικέ μεταφορές στο σύνολο του Βέρλαντ. Έχουμε για παράδειγμα με αυτοκινήτων, ε, ε, μοίρασμένα ποδήλατα, έχουμε τις τοπικές κοινότητες, έχουμε μικρά ε, ηλεκτρικά μηχανάκια ε, και λοιπά. Εάν μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα με διάφορους τέτοιους παράγοντες, ε, μάλλον θα μπορούμε να παρέχουμε πιο καλές και πιο αποτελεσματικές δημόσιες μεταφορές. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup pour votre... Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας με κάποιες καινοτομίες που δεν είχα ακούσει ποτέ μέχρι τώρα αυτή την διάθεση φρέσκων λαχανικών. Απίστευτο μου φαίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Ρόμαν έχει το λόγο για 10 λεπτά. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ ε, στο ε, ενοποιημένο σύστημα δημοσίων μεταφορών ε, στην κεντρική βοημία γύρω από την πρωτεύουσα την Πράγα. Αυτό συμβαίνει με στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες μεταφορών και η παρουσίασή μου είναι χωρισμένη σε διάφορα τμήματα. Πιστεύω ότι είναι ότι υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία εδώ πέρα. Καταρχάς, εδαφικότητα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον περιφερειακό σχεδιασμό. Υποδομές σε μεταφορών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για να έχουμε αποτελεσματικά συστήματα. Ε, αναφέρομαι κυρίως στη, στη υποδομή. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος ε, των τρένων, διότι ε, ε, έχουν πολύ λίγες εκπομπές. Επίσης, μας ενδιαφέρει η σύνδεση με την περαιτέρω περιοχή, με την ευρύτερη περιοχή, την σχέση το ε, ε, ολοκληρωμένο ε, σύστημα δημοσίων μεταφορών και τη σχέση του με τις ατομικές μεταφορές. Και τέλος, θα σας κάνω μία σύντομη σύνοψη και θα σας παρουσιάσω κάποιες συστάσεις. Πώς έχει η κατάσταση. Βρισκόμαστε πράγματι στο κέντρο της Υπήρου της Ευρώπης. Η κεντρική βοημία βρίσκεται ε, στο κέντρο της ε, Τσεχίας είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια στο σύνολο της ε, Τσεχίας. Και από την πτώση του σύντριμου παραπέσματος έχουμε... σημαντική κινητικότητα, το 30% του πληθυσμού μετακινείται προς την Πράγα που αποτελεί σημαντικό κέντρο για τις για την επαγγελματική τους ζωή. Οι υποδομές δεν ήταν αρκετά καλά προετοιμασμένες για την εξέλιξη αυτή και σήμερα ασχολούμαστε ακόμη με τον εξυγχρονισμό και την διεύρυνση των υποδομών για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στη ζήτηση. διοικητική κατανομή μέχρι το 2000 η περιφέρεια ήταν χωρισμένη σε 12 σε 12 δήμους και τώρα έχει αρθεί αυτό. Έχουμε λοιπόν τώρα την κεντρική βοημία και στο κέντρο της βρίσκεται η πρωτεύουσα η Πράγα. Αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα της κεντρικής βοημίας, ε, διότι η έδρα των ε, αρμοδίων φορέων βρίσκεται στην Πράγα. Είναι η μεγαλύτερη από τις περιφέρειες της Τσεχίας, 1,4 εκατομμύρια ε, κατοίκους έχει σχεδόν ε, και η έκτασή της είναι 11.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. επειδή αντικαταστάθηκαν ε, οι νομαρχίες από μία μεγάλη ε, περιφέρεια, Έχουμε μεγάλους δήμους με διευρυμένες αρμοδιότητες, το οποίο σημαίνει ότι οι τοπικές αρχές βρίσκονται έτσι πιο κοντά στους πολίτες και ότι δεν πρέπει απαραίτητα να πάει κανείς στην πρωτεύουσα για να κάνει τη δουλειά του. Οι αποστάσεις ε, λοιπόν έχουν μειωθεί που πρέπει να διανύσει κανείς ε, διότι ε, πολλά πράγματα ρυθμίζονται σε επίπεδο Δήμου. Δυτικά της Πράγας έχουμε την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή, ενώ η πιο αραιοκατοικημένη είναι στην πόλη Ρακόβνικ. Αυτό έχει να κάνει με ε, την ε, μαζική μετανάστευση προς το κέντρο της ε, βοημίας. Όπως σας είπα ήδη, εκεί βρίσκονται οι καλύτερες θέσεις απασχόλησης, οι καλύτερες ευκαιρίες να βρει κανείς ε, καλή δουλειά, ενώ το Ράκοβνικ ε, παραμένει στην περιφέρεια διότι δεν υπάρχουν ε, καλές συνδέσεις με την Πράγα. Μόνο με λεωφορείο μπορεί να πάει κανείς ή με το αυτοκίνητο. Το Ρακόβνικ λοιπόν παραμένει αποκλεισμένο από την μαζική ανάπτυξη. Οδικές ε, υποδομές. Δεν ξέρω αν βλέπετε καλά το διάγραμμα. Με MOV είναι η αυτοκινητόδρομη της κεντρικής βοημίας. Και το Ράκοβνικ βρίσκεται και εδώ στη χειρότερη θέση. Πολύ μικρό κομμάτι αυτοκινητόδρομου οδηγεί προς ε, το Ρακοβνίκ. Ε, είναι λοιπόν ε, μειονεκτική η περιοχή αυτή και όχι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. 70 χιλιόμετρα χωρίζουν το Ράκοβνικ από την Πράγα. είναι μια απόσταση την οποία μπορεί να διανύει κανείς κάθε μέρα για να πάει στην πρωτεύουσα, αλλά αυτό προϋποθέτει ε, σιδηρόδρομο. Εάν υπάρχουν καλοί σιδηρόδρομοι, ε, μπορεί κανείς ε, να διανύει και 130 χιλιόμετρα για να πάει στη δουλειά του. Όσον αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο, υπάρχουν ενιαίες τιμές στην Πράγα και την Κεντρική Βοημία. Οι άνθρωποι λοιπόν χρειάζονται ένα εισιτήριο μόνο και μπορούν να ταξιδέψουν με οποιαδήποτε εταιρεία. Επίσης τα εισιτήρια δεν, έχουν, ε, δεν τυπώνονται απαραίτητα σε χαρτί, υπάρχουν έξυπνες κάρτες που εκδίδουν κάποιες από τις εταιρείε ή ο διαχειριστή του συστήματος. Μπορεί κανείς ε, να κατεβάσει εφαρμογή στο τηλέφωνό του. Έχουμε και ε, εικονικά εισιτήρια, τα οποία μπορεί να φορτώσει κανείς σε τραπεζική κάρτα. Οι ταξιδιώτες δεν χρειάζεται να έχουν κάποιο ειδικό μέσο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ό,τι έχουν στα χέρια τους και να φορτώσουν εκεί ένα εισιτήριο η ολοκλήρωση, η ενοποίηση των ε, μεταφορών ε, έχει ελλείψεις ε, στην περιοχή του Ρακόβνικ. Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Από τις 15 Δεκεμβρίου 2019 όμως προβλέπεται η ολοκλήρωση του συστήματος και βλέπετε εδώ στο σχεδιάγραμμα τι προβλέπεται να γίνει σημαντικό για την ε, ολοκλήρωση των μεταφορών ε, είναι ότι αυτές τις ε, γραμμές δεν τις έχει χαράξει η εταιρεία, η ιδιωτική. Είναι κάτι που έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με τους Δήμους και τις κοινότητες. Έχουν συζητήσει οι Δήμοι και οι κοινότητες με τους πολίτες τους και έτσι έχει διαπιστωθεί που υπάρχουν ανάγκες και τι συχνότητα μεταφορών απαιτείται τι ανάγκε υπάρχουν λοιπόν, ε, πότε πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, πότε πάει κανεί ε, στη δουλειά του. Αφενό αυτό λοιπόν, ενώ από την άλλη ε, στην πόλη του Ρακόβνικ έχουμε περιφερειακές γραμμές που αποτελούν και τμήμα των αστικών μεταφορών. Μία από τις γραμμές ξεπερνάει τα όρια της πόλης, αλλά με το ίδιο εισιτήριο. Έχουμε λοιπόν ένα ενοποιημένο πρότυπο. Αυτή λοιπόν είναι μία εναλλακτική λύση σε σχέση με την ε, ατομική μεταφορά. Σε αυτό το σχεδιάγραμμα βλέπετε τη σιδηροδρομική γραμμή. Πριν 160 χρόνια κατασκευάστηκε και δεν έχει εξυγχρονιστεί έκτοτε. Δεν ε, έχουν γίνει βελτιώσεις ώστε να επιτρέπεται η χρήση γρήγορων ε, σειρμών. Πρέπει να γίνουν πολλά λοιπόν, ώστε ο σιδηρόδρομος ε, να ωφελεί την περιοχή. Εδώ θέλω να σας δείξω πώς παρεμβαίνει το κράτος ε, στις ε, μαζικές μεταφορές. Όλα αυτά γίνονται με βάση τον κανονισμό 1371 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών Έχουμε την πράξη για τις ε, μαζικές μεταφορές ε, και πρέπει να υπάρχει ένα κρατικό σχέδιο για τις μαζικές μεταφορές ε, και έχουμε ένα τέτοιο το οποίο θα τεθεί σε ισχύ στις 30 Σεπτεμβρίου του 2020. Το κράτος και οι περιφέρειες θα πρέπει να έχουν σχέδιο για τις μαζικές μεταφορές και υπάρχει ένα τέτοιο το οποίο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2012. Επιπλέον θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία και σημαντικό είναι και το θέμα της διαλειτουργικότητας ε, όσον αφορά τα εισιτήρια. Οργανώνονται δημόσιοι διαγωνισμοί ε, και επίσης καθορίζονται τα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας. Ε, επίσης υπάρχει κανόνας σχετικά με την η ηλικία των οχημάτων. Σημαντικές είναι και οι εκτόσεις στα εισιτήρια, παιδιά κάτω των 6 ετών ε, ταξιδεύουν δωρεάν, ε, ενώ μέχρι τα 15 έχουν έκπτωση 75%, ε, όπως και οι φοιτητές και όπως και οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών. Το κράτος αποζημιώνει τις επιχειρήσεις για αυτές τις εκπτώσεις. 70 εκατομμύρια το χρόνο πληρώνονται στις εταιρείες αυτές κάθε χρόνο. Επιπλέον, η περιφέρεια αυτή, επειδή βρίσκεται αρκετά μακριά από την Πράγα, έχει υπογράψει συνθήκη και το κράτος ε, έχει δηλώσει τη διάθεσή του να αναλάβει το κόστος αυτού του 75%. Εδώ βλέπετε τις αποστάσεις από τις διάφορες περιφέρειες μέχρι την Πράγα. Και πολύ ευχαρίστω. Θα σα δώσω περισσότερε εξηγήσει κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Σα ευχαριστώ πολύ και στο συγγνώμη που μακρηγόρησα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Στέρμπα για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή ε, παρουσίαση. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να τηρεί πάντα κανεί το χρόνο αγόρευση και έχετε ιδιαίτερο πάθο βέβαια για τον τομέα σα, άρα δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, τελευταία ομιλία, αλλά εξίσου σημαντική από τον κύριο Κρίστιανσεν. Μπορείτε να μα πείτε, παρακαλώ πολύ, τι γίνεται με αυτή την βελγική πλατφόρμα, την Mobiel 21. Θα μα τα πείτε όλα. Περιμένουμε από εσά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε καταρχάς για την πρόσκλησή σας. Θα ήθελα σήμερα να μου επιτρέψετε να σας παραθέσω εδώ την εμπειρία ενός χρήστη των χρηστών εκείνων που χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Καταρχάς, ας κάνουμε μία μικρή άσκηση. Φανταστείτε ότι θα πρέπει να αρνηθείτε μία νέα θέση απασχόλησης, μία δραστηριότητα αναψυχής, ένα πρόγραμμα κατάρτισης εκπαίδευσης, μόνο και μόνο επειδή δεν μπορείτε να πάτε μέχρι εκεί. Με αυτήν είναι η καθημερινότητα όλο και περισσότερων ανθρώπων. Αυτό αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτε στην καθημερινότητά του και αυτό καταδεικνύουν πάρα πολλέ έρευνε και μελέτε που έχουν γίνει σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι ιδιαίτερα θλιβερό. Στο πολύ όμορφο αυτό οικοδόμημα το οποίο ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά επέσχυντο τη σήμερον ημέρα να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξέρετε ότι μιλάμε όλο και περισσότερο για βιώσιμη κινητικότητα. Πάρα πολλά ωραία κείμενα τα οποία μα λένε ότι η κινητικότητα αυτή δεν θα πρέπει απλώ να είναι ασφαλή, οικολογική, οικονομικά προσιτή και προσβάσιμη, αλλά και δίκαιη. Το δίκαιη σημαίνει προσβάσιμη και προσιτή σε όλου. Και ακριβώς ε, σε αυτό έγκυται η λεγόμενη ένδυα όσον αφορά την κινητικότητα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, που πρέπει να αρνηθούν κάποιες ευκαιρίες μόνο και μόνο που δεν μπορούν να μεταβούν στον τόπο που πρέπει να πάνε. Πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν αυτοκίνητο, επειδή δεν έχουν πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες λόγω της ηλικία, λόγω της αναπηρίας τους ή λόγω του τόπου κατοικίας τους. Και ακριβώς αυτό εστιαζόμαστε σήμερα στις αεροκατοικημένες εκείνες περιοχές όπου πάρα πολλοί άνθρωποι πραγματικά είναι εγκλωβισμένοι επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν αυτοκίνητο και δεν είναι διαθέσιμες οι απαραίτητες δημόσιες συγκοινωνίες. 16,7% αυτό είναι το ποσοστό των ανθρώπων που κινδυνεύουν από χαμηλό εισόδημα. Συμφωνώ μαζί σας ότι ο δείκτης αυτός δεν είναι ο πλέον κατάλληλος δείκτης όσον αφορά την ένδυα στα πλαίσια της κινητικότητας, αλλά είναι ένας πολύ καλός δείκτης, τουλάχιστον μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε περισσότερο το ζήτημα αυτό της κινητικότητας και της ένδυας. 16,7% το ποσοστό αυτό δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Η φτώχεια η ένδυα, και επανέρχομαι σε αυτό, είναι ένα ολόκληρο δίκτυο κοινωνικού αποκλεισμού. Σαν τον ιστό που βλέπετε στην φωτογραφία αυτή τη στιγμή. Η έλλειψη κινητικότητας είναι η κόκκινη κλωστή ε, σε αυτό το δίκτυο κοινωνικού αποκλεισμού. 150 κοινωνικά αισθητούτα συμμετείχαν σε μία μελέτη και ασχολούνται με τους φτωχούς και μολονότι η κινητικότητα δεν αποτελεί ένα κεντρικό θέμα το οποίο μελετάνε, παρόλα αυτά τα αισθητούτα αυτά αντιμετώπιση φτώχειας έχουν δει ότι οι περισσότεροι άποροι πλήττονται κατά 90% και από το ζήτημα της ένδυα στην κινητικότητα, το γεγονό ότι δεν μπορούν να πάρουν δημόσιε συγκοινωνίε. Βλέπουμε ότι η έλλειψη κινητικότητα οδηγεί στο κοινωνικό αποκλεισμό και βλέπουμε ακόμα και ότι οι φτωχοί, και το λέω κάπως σωμά, οι φτωχοί ταξιδεύουν λιγότερο. Οι φτωχοί, οι άποροι ταξιδεύουν σαφώς πολύ λιγότερο από ότι εμείς. Και μια αισιόδοξη βέβαια παρατήρηση είναι ότι οι φτωχοί ταξιδεύουν με τρόπο πιο οικολογικό, πιο φιλοπεριβαλλοντικό, πιο πράσινο. Αυτό δεν αποτελεί συνειδητή επιλογή, αλλά μια αναγκαιότητα. Δεν έχουν καμιά άλλη επιλογή ουσιαστικά. Τώρα, Ποιοι είναι οι πιο δύσκολα προσβάσιμοι προορισμοί. Πρώτα απ' όλα βλέπετε τον τόπο εργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για του ανθρώπου αυτού να έχουν πρόσβαση στον τόπο εργασία. Στη δεύτερη και τρίτη θέση βλέπουμε τον τόπο που ζει η οικογένειά του, του φίλου, τι δραστηριότητε τη αναψυχή, την νομική περίθαλψη, αλλά ακόμα και τα προγράμματα κατάρτιση και τα προγράμματα εκπαίδευση, τα οποία δεν καταφέρνουν να έχουν πρόσβαση. Α δούμε ένα παράδειγμα από την αγορά εργασία στην Φλάνδρα, στην περιφέρεια του Λίνμπορκ. Πραγματικά μου προκάλεσαν εντύπωση τα δεδομένα αυτά. Λιγότερο του 20% των θέσεων απασχόληση, οι οποίε απαιτούν μία ώρα οδήγηση, είναι προσβάσιμες εξίσου σε μία ώρα με δημόσιε συγκοινωνίε σε, καταλαβαίνετε ότι είναι επέσχυντο αυτό για μια περιφέρεια σαν τη Φλάνδρα, η οποία είναι πυκνοκατοικημένη. Δεν τολμώ να φανταστώ ότι μπορεί να συμβαίνει σε αεροκατοικημένε περιοχέ. Επίση, το δίπλωμα οδήγηση αποτελεί πλέον απαιτούμενο επαγγελματικό προσόν. Πολύ συχνά οι άνθρωποι δεν καταφέρουν να αποκτήσουν μια θέση απασχόληση επειδή δεν έχουν το δίπλωμα οδήγηση. Ένα ακόμα πολύ θλιβερό αποτέλεσμα από τη μελέτη αυτή είναι ότι το να αναζητήσει κανεί θέση απασχόληση χωρί αυτοκίνητο απαιτεί έξι μήνε παραπάνω αναζήτηση. Και επίση βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι στην αναζήτηση θέση απασχόληση το μορφωτικό επίπεδο δεν είναι πλέον ο πιο καθοριστικό παράγοντα. Ο πιο καθοριστικό παράγοντα είναι η προσβασιμότητα. Ο τρόπο που μεταβαίνει κανεί προ αυτόν τον τρόπο εργασία. Πριν τη μελέτη αυτή, πριν τη διαβάσω, πριν γνωρίσω τα πορίσματά τη, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσε να ισχύει ή κάτι τέτοιο. Ποια είναι όμω τα πραγματικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα κινητικότητάς μα. Καταρχά και θα σα κάνει εντύπωση αυτό, είναι η έλλειψη χρηματοοικονομικών πόρων. Αλλά πολύ συχνά δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα μεταφορά. δεν υπάρχουν τα αυτοκίνητα, δεν υπάρχουν κοντά στάσει λεωφορείων, οι συνδέσει είναι πολύ κακέ. φυσικοί περιορισμοί, έλλειψη επίση δεξιοτήτων. Δεν μπορώ να διαβάσω, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω πώ λειτουργεί το δημόσιο σύστημα μεταφορών. Επίσης, σε περιοχές όπως η Φλάνδρα, ακόμα 50.000 άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν ποδήλατο. Αυτό είναι ασύλληπτο για μένα που ζω στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν και ψυχολογικά εμπόδια, ο φόβος το να πάρει κανείς τις δημόσιες κοινωνίε. Από τη Λουβέν, 12 λεπτά με το τρένο, απέχει μία πόλη και πολύ πολίτες φοβούνται να μπουν στο τρένο αυτό και να, πούνε, να πάνε στο γειτονικό αυτό προάστιο. Γιατί πολλοί φοβούνται ότι μπορούν να καταλήξουν στι Βρυξέλλες και τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή. Υπάρχουν και γνωστικά εμπόδια. Επίση, δεν υπάρχουν απαραίτητε υποδομέ, δεν υπάρχει απαραίτητη ενημέρωση. Υπάρχει επίση διακριτική μεταχείριση. Και αυτό πολλέ φορέ μπορεί να λειτουργήσει ω εμπόδιο για την κινητικότητα. Τώρα, όταν μιλήσαμε με αυτά τα 150 Ινστιτούτα αντιμετώπιση τη φτώχεια μα είπαν ότι οι βασικοί παράγοντε καταρχά που συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτή τη μειωμένη κινητικότητα είναι καταρχά ότι έχουμε να κάνουμε κυρίω με πολίτε οι οποίοι δεν εργάζονται τι συνήθει ώρε εργασία. Πρέπει να φύγουν για παράδειγμα στι 5 η ώρα το πρωί, επομένω δεν έχουν δημόσιε συγκοινωνίε εκείνη την ώρα. Στη Φλάνδρα κατά μέσο όρο οι δημόσιε συγκοινωνίε ξεκινάνε κατά τι 7 ή τι 8 το πρωί. Επίση, το κόστο θα πρέπει να είναι προσβάσιμες αυτέ οι Ξέρετε ότι στο Βέλγιο δικαιούται κανείς ένα είδος αποζημίωσης. Αυτό άκουσα και από τον Τσέχο συνάδελφο. Μα θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό κανείς και για να το γνωρίζει θα πρέπει να το ρωτήσει. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, ένα αυτόματο δικαίωμα στην αποζημίωση αυτή. Δεν χρειάζεται κανείς να ετηθεί την αποζημίωση αυτή, θα πρέπει να του δίδεται αυτόματα. Επίσης, ε, ενημέρωση για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δημόσιες συγκοινωνίε μας. Η κινητικότητα μπορεί να αποτελήσει μια λύση, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχουν και απαραίτητες πληροφορίες ή απαραίτητη ενημέρωση. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μόνο για παράδειγμα μέσω ενός έξυπνου τηλεφώνου. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν έχουν πρόσβαση σε ένα έξυπνο ευφυές τηλέφωνο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι πληροφορίες αυτές να διατίθενται πολύ εύκολα και εκτός διαδικτύου, εκτός έξυπνων συσκευών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύπλοκο το πρόβλημα αυτό της ένδυας και της κινητικότητας. Μπορούμε να έχουμε βέβαια κάποια λύση στο πρόβλημα αυτό. Ξέρετε ότι ε, ακούγονται Πολλέ ιδέε που έχουν να κάνουν με τη λεγόμενη συμμετοχική επιμερισμένη κινητικότητα. Μπορεί όμω αυτή από μόνη τη να αποτελέσει λύση. Δεν νομίζω, μια μερική μόνο λύση, γιατί για να χρησιμοποιηθούν οι κοινέ αυτέ οι υπηρεσίες χρειάζονται δεξιότητε προσβασιμότητα, χρειάζονται πιστοτικέ κάρτε. Έχουμε και το ψηφιακό χάσμα, η πληροφορία η ενημέρωση είναι αρκετά κατακαιρματισμένη. στι Βρυξέλλε, για παράδειγμα, η ενημέρωση για τα διάφορα συστήματα επιμερισμένη κινητικότητα είναι αρκετά κατακαιρματισμένη ή δυσέβρετη στο ίδιο το δίκτυο προσφορά τέτοιων συγκοινωνιών είναι αρκετά περιορισμένη. Τι έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε εμείς. Συμμετέχουμε σε διάφορα project, σε διάφορα προγράμματα και βλέπετε εδώ πέρα ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, οι βασικοί φορείς. Για παράδειγμα, βλέπετε εδώ πέρα ότι δεν εκπροσωπούνται οι ομάδε χαμηλού εισοδήματο. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν διαβάζουν, και επίση, δεν συμμετέχουν, δεν βρίσκονται στον κατάλογο αυτό. Ως κοινότητες λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το ζήτημα αυτό για να καταφέρουμε να εντάξουμε περισσότερο και αυτές τις πιο ευάλωτες ομάδες. Και τι μπορούμε να κάνουμε. Να εμπλέξουμε αυτές τις ευάλωτες ομάδες στις συναντήσεις που κάνουμε. Κάθε φορά που μιλάμε για τα βιώσιμα σχέδια αστικής κινητικότητας θα πρέπει και αυτοί να μπορούν να συμμετέχουν. Θα πρέπει να μπορούν να συνεργαστούμε μαζί τους, να μιλάμε τη γλώσσα τους. Ξέρετε ότι το πρόβλημα αυτό της κυκλοφοριακής ένδυας είναι πολύ πλοκό πρόβλημα, πολύ σχηδές, πρέπει να βρεθούν πολύ, πολλές διαφορετικές λύσεις και θα πρέπει να εμπλακούν διάφοροι, διάφορες πολιτικές. Η πολιτική της, των ίσων ευκαιριών, η πολιτική της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και πολλές άλλες κοινωνικές πολιτικές μπορούν να συμβάλλουν από κοινού στο να επιληθεί το ακαθόδες αυτό πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ αυτή η τελευταία παρέμβαση μας κάνει κάπως να παγώνουμε γιατί είμαστε το 2020 και υπάρχουν ακόμη πάρα πολλοί άνθρωποι. Ξέρετε, μιλάμε για ενεργειακή φτώχεια. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν θέρμανση στο σπίτι τους ή δαπανούν το 1 τέταρτο του μισθού τους για να πληρώνουν λογαριασμούς ενέργειας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να εργαστούμε και για αυτό το θέμα του επισφαλούς στις μεταφορές. Και θα πρέπει να παρουσιάζονται και στα κείμενα και στα θεσμικά όργανα. Και ενώ θεσπίζουμε πλατφόρμες για την καταπολέμηση της ανέχειας και είπατε κάτι εξαιρετικά στην ε, εισαγωγή σας θα θέλανε οι άνθρωποι αυτοί να βρουν δουλειά, έχουν τις ικανότητες αλλά δεν μπορούν γιατί δεν έχουν τα μέσα για να μπορούν να μετακινηθούν. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ο πίνακας αυτός. Ας περάσουμε κατευθείαν στη συζήτηση. Λοιπόν, κύριε Ντάνιλσον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Ε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονε για τις παρουσιάσεις τους. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι διαφορετικέ προοπτικέ σας. Διότι αν θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε τον τομέα των μεταφορών ε, θα πρέπει να φροντίσουμε, να προσαρμόσουμε τις μαζικές μεταφορές ε, σε όλους τους ανθρώπους. Και έχω κάποιες ερωτήσεις προς εσάς. Καταρχάς, ε, σύμφωνα με τις δικές σας εμπειρίες, ε, ποια είναι τα σημαντικότερα εμπόδια για την εξέβρεση καινοτόμων λύσεων για τις ε, συλλογικές μεταφορές, τις μαζικές μεταφορές. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η χρηματοδότηση από το δημόσιο. Μας λείπουν δηλαδή οι καινοτόμες λύσεις ή μας λείπουν οι πόροι, η χρηματοδότηση. Και μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Μια και βρίσκεστε εδώ και μας παρουσιάζετε τις διάφορες περιπτώσεις σας εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι περιμένετε εσείς από εμά, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε στις περιφέρειες σας. Και τρίτον, και ο Ματίας το ανέφερε αυτό το θέμα της, των μαζικών μεταφορών κατόπιν ζήτησης. Υπηρεσίες που παραγγέλνει κανείς κατά περίπτωση. και πώς μπορούμε να ε, ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο ε, εκτείναξης του κόστους. Και τέταρτον, σε σχέση με το ε, παράδειγμα της ε, Πορτογαλίας. Ε, υπάρχουν αεροκατοικημένες περιοχές όπου μπορεί κανείς να πάει σε μεγάλη πόλη διανύοντας μικρότερη απόσταση, περνώντας τα σύνορα. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει κάτι. Πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τέτοιες διασυνοριακές μαζικές μεταφορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντάνελσον. Κυρία Αρμάν. Ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οι περισσότερες αναπτυγμένες χώρες ε, ε, έχουν ε, εγκαταλείψει την εξοχή και στις φτωχές χώρες αν πρέπει κάποιος να έχει έναν καλό μισθό πρέπει να πάει στις πόλεις. Στη Ρουμανία από που προέρχομαι έχουμε το 40% του πληθυσμού και παραπάνω να ζει στην υπεθρό. Λέμε ότι καλό είναι αυτό, είναι βιώσιμο, όμως ε, στην πραγματικότητα ε, επιδίδονται σε μία γεωργία επιβίωσης. Βέβαια, αυτό ξεπερνά το 16,7% που αναφέρεται. Μιλάμε για 40% και οι άνθρωποι αυτοί μετακινούνται ε, ένα μέρος και με κάρα μάλιστα. Ε, Εμεί θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια οικονομία με χαμηλό άνθρακα και θέλουμε να διατηρήσουμε και αυτό τον ε, χαρακτήρα τη υπαίθρου. Μας ε, λένε ότι αυτό είναι πλέον έκτημα, όμως πώς θα λύσουμε αυτή την εξίσωση, γνωρίζοντα πως αν 30-40 χρόνια πριν υπήρχε σε όλα αυτά τα χωριά το τρένο, σήμερα δεν υπάρχει πια και το χάρη, αν μια χώρα όπως, την, ε, όπως η Γαλλία δυσκολεύεται να συνδέσει τα χωριά με σιδηρόδρομο, σκεφτείτε τι συμβαίνει στη Ρουμανία, ε, που τα τρένα δεν κυκλοφορούν ε, καν στις βασικές διαδρομές μεταξύ των μεγάλων πόλεων. Έτσι λοιπόν, ε, πώς ε, συνεχίζουμε να προστατεύουμε ε, αυτή τη ζωή στην Ήπεθρο που συνεχίζει να υπάρχει σε κάποιες χώρες. Θα συνεχίσουμε να την προστατεύσουμε ή θα ακολουθήσουμε την ίδια οδό με τις αναπτυσσόμενες χώρες, με τις αναπτυγμένες χώρες, συγγνώμη. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν από την Ήπεθρο και πήγαν στις πόλεις. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια επαλλογή. Θα ακολουθήσουν αυτές οι χώρες την ίδια οδό που ακολούθησε και η Δύση. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε για αυτόν τον προβληματισμό, κύριε Άρβο. Θα το ξανασυζητήσουμε. Θα σας απαντήσουν οι εμπειρογνώμενες. Ο κύριος Ολιβιέ. Ναι, εγώ θέλω να συνεχίσω τόσο είπε και συνάδελφος. Σίγουρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την αδικία που υπάρχει ε, για τους ανθρώπους που ζουν σε αεροκατοικημένες περιοχές. Ε, έχουμε ακούσει πολλά όμως ε, εγώ βλέπω ότι υπάρχουν ε, λίγες λύσεις. Πάντοτε καλό είναι να συμμετέχουν ε, οι πολίτες και να ζητάμε τη γνώμη τους, όμως δεν καταλαβαίνω πώς οι εμπειρογνώμονες ή οι πολίτες θα μπορούσαν να βρουν λύσεις σε γιγάντια προβλήματα. Ας δούμε την προσφορά. Τότε θα δούμε ότι είναι γνωστές οι προσφορές, το τρένο, το μοίρασμα του ΙΟΤΑΧΗ και τα λοιπά. Ε, στην Αφρική έχουμε και συλλογικά ε, ταξί, παύλα λεωφορεία που εξυπηρετούν τις ανάγκες αλλά παρόλα αυτά ε, είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες αυτές. Η θεμελιώδης ερώτηση είναι επιλογή της κοινωνίας, δηλαδή αν θα συνεχίσουμε την αστικοποίηση και αν όλα θα τα ομαδοποιήσουμε και θα τα συγκεντρώσουμε σε πολύ μικρούς ε, χώρους, στο σύνολο των δραστηριοτήτων. Η απάντηση λοιπόν ε, σε αυτή την αδικία ίσως ε, δεν αφορά το θέμα της κινητικότητα, αλλά τη χωροταξία. Δηλαδή να έχουμε πιο εναρμονισμένε επικράτειες ε, και να έχουμε υπηρεσίες που θα προσφέρονται στους ανθρώπους και να προσφέρονται και πολιτιστικές δραστηριότητες στους ανθρώπους αυτού παρά να τους καλούμε κάθε μέρα να φεύγουν και να κάνουν χιλιόμετρα για να πάνε στο σινεμά, στο θέατρο, στη δουλειά τους. Μιλάμε λοιπόν ε, για τεχνικές και για τρόπους μεταφοράς, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε όμως για κοινωνικά μοντέλα. Ευχαριστώ κύριε Ολιβιέ, η κυρία Ντεπερνέ. Ευχαριστώ και εγώ για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα και πραγματικά σας ευχαριστούμε για το πώς παρουσιάσατε το πρόβλημα. Εγώ συμμετέχω στην Επιτροπή Μεταφορών αλλά και στην Επιτροπή Γεωργίας ε, και ε, τη ανάπτυξη ε, τη Επέθρου περιφερειακή ανάπτυξη. και βλέπουμε ότι συνδέονται όλα αυτά τα θέματα, δηλαδή ακριβώ πώ αναπτύσσεται η Επέθρο, που είναι συνήθω η πιο αραιοκατοικημένη και πώ θα επιτρέψουμε στου πολίτε και σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο να συμμετέχουν στην κινητικότητα. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν μπορούμε να βγούμε από τα στεγανά, το πρόβλημά πρόβλημά είναι ότι δεν μπορούμε να βρούμε τα στεγανά. Ε, δηλαδή, σε μια επιτροπή μπορούμε να συζητάμε ε, για ε, τις δουλειές στις πόλεις και σε άλλη επιτροπή μιλάμε για τη γεωργία που θα βλάπτει λιγότερο το περιβάλλον. Όμως πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά συνολικά. Η γεωργία σήμερα ε, συνδέεται πάρα πολύ με χημικά προϊόντα ε, και δεν χρειάζεται ε, μεγάλο εργοτικό δυναμικό. Αυτό το ήθελε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι καλούμαστε να ακολουθήσουμε μια άλλη οδό και ίσως θα πρέπει να υπάρξει νέα δημιουργικότητα στη Γεωργία και θα πρέπει η Ήπεθρος να ξαναγίνει ελκυστική και να υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης. Εγώ ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτά τα θέματα ε, και είναι κρίμα γιατί παράλληλα σήμερα το απόγευμα γίνεται μια συζήτηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για το θέμα του Ταμείου Δικής Μετάβασης. Πώς εμείς δηλαδή θα επιτρέψουμε στην αγροτική ανάπτυξη να έχει δίκαιη μετάβαση και εδώ σε στεγανά μιλάμε για τις μεταφορές. Θα πρέπει λοιπόν ε, να σκεφτούμε με έναν ε, πιο ε, εκάρσιο τρόπο και σε επίπεδο δικτύων, σε ψηφιακό επίπεδο, δηλαδή και για τους ανθρώπους που δεν συμμετέχουν σε ψηφιακά δίκτυο, δίκτυα. είδαμε παραδείγματος χάρη το σουηδικό παράδειγμα, δηλαδή μπορεί παραδείγματος χάρη κάποιοι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν. Νομίζω ότι δώσατε και καλά παραδείγματα και πάντοτε υπάρχουν τα διλήμματα, θα πάρω το αυτοκίνητό μου, να πάω για ψώνια κτλ. Εσείς παρουσιάσατε κάποιες λύσεις. Υπάρχουν πολλά θετικά παραδείγματα παντού και πρέπει να κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση του χρητικού κόσμου και να το σκεφτούμε αυτό από κοινού με την κινητικότητα. Ευχαριστώ κυρία Κουντουρά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το ζήτημα της ε, προσβασιμότητας των αρεοκατοικημένων περιοχών έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη, γιατί η ύπεθρο, οι ορεινές, οι νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζουν όλο ένα και πιο έντονα το δημογραφικό πρόβλημα, παρόλο που έχουν κρίσιμο ρόλο για την επισητιστική ασφάλεια, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον τουρισμό, αλλά και για τη γεωστρατηγική της Υπήρου μας. Εν ώψη λοιπόν της πράσινης μετάβασης, τα αστικά κέντρα θα δεχθούν ισχυρές πιέσεις, οι οποίες μπορούν να μειωθούν μόνο αν δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να επιστρέψουν οι κάτοικοι στην περιφέρεια. Η ιστορική συγκυρία, κυρίως λόγω της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας, είναι ευνοϊκή. Γιατί αν το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να δούμε τις μεταφορές στις αεροκατοικημένες περιοχές από μία άλλη οπτική είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο δεν μπορεί να αφαιθεί στους νόμους της ελεύθερης αγοράς γιατί απλά δεν θα επιβιώσει με οικονομικούς όρους. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους ώστε η κοινωνία ο σύνολο να στηρίξει τις απομονωμένες περιοχές της Ευρώπης. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τους εμπειρογνώμονες ποια συγκεκριμένα μέτρα θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια προγράμματα και χρηματοδότηση χρειάζονται στο πλαίσιο της νέας πράσινης συμφωνίας και αν αρκούν τα παραδοσιακά εργαλεία ή ίσως χρειάζεται να, είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των περιοχών αυτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ κυρία Κουντούρα. Κύριο Βιτανόφ, τώρα έχει το λόγο, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω βουλγαρικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Βλέπουμε για ακόμα μία φορά ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες μπορούν να δραματίσουν σημαντικότατο κοινωνικό ρόλο. Πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο λοιπόν την κοινωνική διάσταση των μεταφορών. Οι μεταφορέ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελούν μόνο επιχειρηματική δραστηριότητα. Ιδίω οι δημόσιοι κοινωνίε θα πρέπει να λειτουργούν για του πολίτε και προ το συμφέρον των πολιτών. Δεν θα πρέπει να έχουμε ω μέλημά μα εδώ πέρα την κερδοφορία. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε την απερίμωση των αγροτικών περιοχών, των περιοχών τη υπαίθρου και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε τελικά να δημιουργήσουμε συνδέσμου μεταφορικού με τι περιοχέ περιοχές αυτές. Ως κοιόδης εισηγητής για τον σχετικό κανονισμό θα ήθελα πραγματικά οι συμβάσεις, οι δημόσιες συμβάσεις για τις δημόσιες συγκοινωνίες να προστατευθούν και να μπορούμε να διασφαλίσουμε τις συγκοινωνίες αυτές ακόμα και όταν δεν θεωρούνται, δεν αξιολογούνται ως επικερδείς. Ξέρετε ότι αν ακολουθήσουμε εδώ πέρα ως γνώμονα μόνο το ιδιωτικό κέρδος, τότε σίγουρα οι α, περιφερειακές συγκοινωνίες οι οποίες ε, εξορισμού δεν είναι επικερδείς, σιγά σιγά θα εξαφανιστούν. Θα πρέπει επίσης ε, να λάβουμε υπόψη μας τα βασικά δικαιώματα στην κινητικότητα όλων των πολιτών. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα των δημοσίων συγκοινωνιών και να αποφύγουμε σε κάθε περίπτωση την ιδιωτικοποίησή τους. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Βιτανόφ. Όντως τίθεται ένα σημαντικό το ζήτημα όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων συγκοινωνιών. Είναι ένα πραγματικό ζήτημα αυτό το οποίο θέτεται αυτή τη στιγμή για την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων συγκοινωνιών και ξέρουμε ότι σε πάρα πολλές πόλεις Ευρώπης η τάση αυτή έχει προκαλέσει πρόβλημα. Η κυρία Κουντουζά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και ιδιαίτερα για τη δική μας ε, πολιτική οικογένεια, αλλά και όλοι μας ε, θα πρέπει να πιστέψουμε ότι αν θέλουμε πραγματική αλλαγή στην πολιτική, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, να παραβλέψουμε καμία περιφέρεια, καμία περιοχή. Και εγώ προέρχομαι από το μικρότερο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Μάλτα, και μάλιστα από το μικρό ε, νησί του Γκότζο, που δεν είναι το βασικό νησί της Μάλτας. Και ενώ έχουμε αρκετά καλές διασυνδέσεις ε, με τις ε, διάφορες περιοχές, ε, αντιμετωπίζουμε την απομόνωση και τα προβλήματα που συνδέονται με αυτήν. Βλέπουμε διαφυγή επιστημόνων, πολύ πάνε να δουλέψουν στο βασικό νησί, το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Παρ' αυτά πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες και πιο κοντά ε, στο σπίτι του καθενός. Ε, και όλα αυτά επηρεάζουν και τη ζωή μας, ε, διότι υπάρχουν ζευγάρια που μετακομίζουν στο μεγάλο νησί, διότι παρότι είναι καλές οι συνδέσεις, προτιμούν να μετακομίσουν. Και θέλω να σας εξηγήσω λίγο την κατάσταση, διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αεροκατοικημένες περιοχές είναι ακόμη μεγαλύτερη υποχρέωση να δώσουμε καλές ε, συνδέσεις, ε, καλές μεταφορές στους ανθρώπους αυτούς. Αλλιώς ε, η ελεύθερη κινητικότητα που είναι τόσο θεμελιώδης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ισχύει για τις περιοχές αυτές και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου αυτόν τον στόχο, διότι ακόμη και αν είναι δύσκολο, διότι ο ιδιωτικό τομέα δεν θέλει να επενδύσει σε αυτέ τι απόμακρε περιοχέ, οι δημόσιε αρχέ πιστεύω ότι έχουν ευθύνη να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς να τους δώσουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό ή ε, σε άλλα μέρη του ιδίου κράτους μέλους για να έχουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, ε, καλύτερες ε, κοινωνικές ε, ευκαιρίες, ε, πολιτιστικές προσφορές. Και άλλωστε οι καλύτερες ε, διασυνδέσεις μπορεί να προσελκύσουν και περισσότερες επενδύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε όλες τις μας περιφέρειες ασχέτως μεγέθους. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουτουζάρα. Και ένα ερώτημα και από μένα τώρα μας παρουσιάσετε διαφορετικές πτυχές των δημοσίων συγκοινωνιών και μας είπατε ότι απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο από τον λεγόμενο αγροτικό κόσμο, τις αγροτικές περιοχές. Μα πρόκειται για μια καθαρή συνειδητή πολιτική επιλογή. Και εκεί πέρα βλέπουμε ότι το ζήτημα όχι μόνο της αστικοποίησης, αλλά και της διακυβέρνηση είναι καθοριστική σημασίας. Και το λέω αυτό διότι όταν επιλέγει κανείς να επενδύσει μόνο για παράδειγμα στο TGV, στα τρένα υψηλή ταχύτητο. Πολύ ωραία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχουν ολόκληρε περιοχέ οι οποίε αποκλείονται. Τα μικρά τρένα τα οποία εξυπηρετούσαν επιμέρου μικρότερε περιοχέ εξαφανίζονται. Άρα θα πρέπει να ταινίσουμε το μέλλον, αλλά με λύσει πιο βιώσιμε, οι οποίε θεωρώ ότι υφίστανται. Παντού στην Ευρώπη υφίστανται βέλτιστε πρακτικέ. Κανεί, για παράδειγμα, δεν έφερε κάτι και ενδεχομένω να είναι λίγο φιλοσοφικό το ερώτημα αυτό. Το θα μπορούσαν να είναι πραγματικά δωρεάν, εντελώ δωρεάν οι το προσεγγίσατε κάπως αυτό στις διαφάνειές σας, διαφορετική διαβάθμιση των θυμών με βάση την ηλικία, αλλά για παράδειγμα στη Γαλλία έχουμε πειραματιστεί με το ζήτημα αυτό και μάλιστα στη Δουνκέρκη έγινε ένα τέτοιο πείραμα για 200.000 κατοίκους δωρεάν μεταφορές. Και τι είδαμε τότε, ότι οι πιο φτωχοί άνθρωποι που δαπανούσαν τόσα πολλά χρήματα για να έχουν ένα αυτοκίνητο μπορούν πλέον να πάρουν δωρεάν τις δημόσιες κοινωνίες. Άλλοι που δεν βγαίνουν από το σπίτι τους κινούνται τώρα περισσότερο. Υπάρχουν λοιπόν και άλλα εργαλεία πέρα από αυτά που είπατε. Δεύτερον, Είμαστε Επιτροπή Μεταφορών εδώ. Δεν είμαστε η Επιτροπή Γεωργίας, ούτε η Επιτροπή του Αγροτικού, θέλετε, κόσμου, των αγροτικών περιοχών. Άρα, θα πρέπει να προτείνουμε κάποια εργαλεία προκειμένου να προωθήσουμε την κινητικότητα και στις αγροτικές περιοχές και στις περιοχές της Υπέθρου. Και υπάρχει το χάσμα των γενναίων και υπάρχει απόκληση ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι είναι πιο ηλικιωμένοι και σε αυτούς οι οποίοι είναι γκίγκ, οι δήμονες πληροφορικής και έχουν πάντα στο χέρι τους ένα κινητό τηλέφωνο. Και ξέρετε ότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή διαδικτύου δεν καλύπτουν και όλες τις περιοχές και ενδεχομένω να βρίσκεται κανείς στην Ήπεθρο, αλλά σε μια περιοχή που έχει υψηλή οικονομική ανάπτυξη, ενώ υπάρχουν και άλλες περιοχές Ήπεθρο που είναι πολύ πιο υποβαθμισμένες οικονομικά. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα καταφέρουμε να εμφυσίσουμε οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές και όχι μόνο να καταφέρουμε να τις προσελκύσουμε αυτές προς τις πόλεις, προς τα αστικά κέντρα. Κάποιες πρώτες ιδέες σας έδωσα τώρα και για τη δική μας την Επιτροπή βέβαια, αλλά και για σας και θα θέλαμε να σας ξανακούσουμε τώρα κυρία Τελές σε σχέση με τις παρατηρήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοι. Σας δίνω λοιπόν τώρα το λόγο πάλι για τουλάχιστον, άντε, πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ. Πολλές ήταν οι ερωτήσεις που τέθηκαν και συγκεκριμένα. Νομίζω ότι κάποιε αναφέρονται στην πορτογαλική περίπτωση του κ. Ντάνιελσον, παραδείγματο χάρη. Εγώ πιστεύω ότι από όσα ακούσουμε, αντιλαμβανόμαστε ξεκάθαρα το εξή, ότι θα πρέπει να βλέπουμε τις μεταφορέ ότι ε, ως ένα παράγοντα ε, κοινωνικής συνιστώσεως Είναι ε, ουσιαστικά το δικαίωμα στις μεταφορές κάτι αναφέρονται και αν δεν έχουμε μεταφορές δεν έχουμε δικαιοσύνη και έχουμε πολλά που μας προσφέρει η κοινωνία, την υγεία, τον πολιτισμό κτλ. Όμως στην περίπτωση της Πορτογαλίας, εγώ μόνο για την περίπτωση αυτή μπορώ να μιλήσω γιατί γνωρίζω καλύτερα, ε, γιατί ε, είδαμε ακριβώς ποιες είναι οι αεροκατοικημένες ε, περιοχές όπου οι άνθρωποι δεν έχουν ίσες ευκαιρίες για τις μεταφορές. Έχουμε, παραδείγματο χάρη, τις χερσαίες μεταφορές με τα λεωφορεία. Και θέλω να απαντήσω στην ερώτηση ποιο είναι το πιο μεγάλο εμπόδιο εμείς έχουμε γραμμές ε, που ε, ουσιαστικά ε, είναι κερδοφόρες και άλλες που δεν είναι. Και έχουμε οικονομικό πρόβλημα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό το πρόβλημα στην Πορτογαλία το ίδιο το κράτος ε, ε, στράφηκε προς τους ιδιώτες, ε, όμως οι ιδιώτες δεν μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί σε μια χώρα που έχει τόσο μεγάλες αεροκατοικημένες περιοχές δεν ήταν κερδοφόρο για αυτούς. Έτσι λοιπόν, η λύση ποια είναι ότι ε, θα πρέπει ο δημόσιο τομέα να ασχοληθεί. Εγώ καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να καλυφθούν οι ρεκοντημένε περιοχέ από το δημόσιο τομέα. Ο δημόσιο τομέα θα πρέπει να εργαστεί για το θέμα αυτό. Και στην περίπτωση τη Πορτογαλία, εμεί χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Χρειαζόμαστε πολλά, αλλά πολύ περισσότερη χρηματοδότηση για τι μεταφορέ. Τα χρήματα βέβαια δεν φτάνουν. Δεν αρκεί όμω να δίνονται χρήματα από την Ευρώπη. Ε, δεν αρκεί αυτό, γιατί εμεί φτιάχνουμε και πολλού ποδηλατών ε, σε περιοχές όπου κανένας δεν χρησιμοποιεί το ποδήλατο γιατί σε αεροκρατικές περιοχές όπου είναι ε, ο πληθυσμό μεγάλη ηλικία δεν χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτοί το ποδήλατο όσο και αν θέλουμε αν δεν έχουμε ανθρώπους ε, πιο νέους και πιο ενεργητικούς οι οποίοι αυτοί θα χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο και θα υιοθετήσουν μια νέα κουλτούρα ουσιαστικά κινητικότητας τότε δεν γίνεται. Και έχουμε αυτό το θέμα. Εμεί ξοδεύουμε χρήματα από την Ευρώπη για να φτιάξουμε υποδομέ που δεν θα χρησιμοποιηθούν. Το ίδιο και εδώ. Εμεί ε, θέλουμε να εργαστούμε στο θέμα των μεταφορών. Τελικά δεν υπάρχουν χρήματα για να αγοράσουμε τον εξοπλισμό. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή σας ε, να αναθεωρήσει όλο το θέμα της χρηματοδότησης που δίνεται στην Πορτογαλία λόγου χάρη για την πρόθεση των μεταφορών. Γιατί εντάξει, εστιάζουμε στην καινοτομία και στο περιβαλλοντικό θέμα, όμως ε, πρέπει η εφαρμογή να γίνεται σύμφωνα με όσα είπε και ο Βέλγος συνάδελφος, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν ούτε ίντερνετ ούτε τηλέφωνο. Και πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά πριν από το να δίνονται τα κονδύλια. Πρέπει να γίνονται μελέτες. Γιατί θα πρέπει να έχουμε βιώσιμες οικονομικά λύσεις, όμως θα πρέπει να δούμε και σε ποιες επικράτειες στοχεύουμε. Και πολλές φορές γίνονται δρόμοι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι τους δρόμους αυτούς με τα αυτοκίνητά τους, αλλά ε, τελικά... Ε, οι άνθρωποι επειδή είναι ε, σε πολύ αεροκατοικημένε ε, περιοχές ε, δεν μπορούν να φτάσουν καν στο σπίτι τους. Μπορεί να είναι γεμάτο λακκούβες ο δρόμος, μπορεί να έχει ποτάμια. Επίση δεν μπορεί οποιοδήποτε να περάσει από αυτούς τους δρόμους. Πρέπει να σχεδιαστεί λοιπόν όλο αυτό θα πρέπει να έχουμε και χωροταξία. Όμως, όπως είπε και η Πρόεδρος, εδώ μιλάμε για μεταφορές και κινητικότητα. Και θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό κάθε χρηματοδότηση που δίνεται από την Ευρώπη στην Πορτογαλία να συνοδεύεται από μία μελέτη, από ένα σχέδιο που θα συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους τρόπους μεταφοράς. Γιατί, ε, παραδείγματο χάρη, από το σπίτι του να πάει κάποιο μέχρι το ταχυδρομείο ε, και το αν θα πάει με τα πόδια ή αν θα χρησιμοποιήσει ε, το αυτοκίνητό του ή αν θα πάρει το λεωφορείο. Θα πρέπει η στάση, παραδείγματο χάρη, να είναι καλυμμένες ε, με στέγαστρα ε, οι στάσει γιατί στην Πορτογαλία ούτε ένα παγκάκι δεν έχει να καθίσει κανείς, ε, ούτε ένα δέντρο δεν υπάρχει. Δηλαδή για έναν ηλικιωμένο που είναι μόνο του, τελικά μάλλον θα πάρει το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν μιλώ για μια στρατηγική εδώ. Πριν να ταπανηθούν τα χρήματα πρέπει να σκεφτόμαστε, πρέπει να έχουμε στόχους και στρατηγική και μέθοδο και στόχους και σχεδιασμό. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε φυσικά και τα κοινωνικά μοντέλα. Εγώ ε, φυσικά πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ε, την ίδια επιτυχία όπως ε, βλέπουμε τώρα στις μεγάλες πόλεις όπου υπάρχουν τα πάντα όμως και στην υπηρετική χώρα βλέπουμε μεγάλες αλλαγές και εμείς έχουμε βιολογική γεωργία έχουμε νέους γεωργούς που ζουν στην υπηρετική χώρα, στο κέντρο της χώρας και Επίσης ε, τα πορτογαλικά ε, μιλούνται και παντού στον κόσμο. Δεν ε, έχουμε μόνο τουρίστες στο Αλγκάρβε, αλλά έχουμε τώρα τουρισμό και στο βόρειο τμήμα της χώρας, ακριβώς γιατί είναι διαφορετικοί οι άνθρωποι εκεί, έχουν ταυτότητα, έχουν εντελώ διαφορετικούς τρόπους ζωής, διαφορετική κουλτούρα και είναι διαφορετικός ο τρόπος που ζουν και ο τουρίστας θέλει να δει αυτή τη διαφορά και μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτή τη διαφορά αν έχουμε φυσικά πιο ευέλικτες μεταφορές, σε πιο μικρή κλίμακα. Ε, γιατί μπορούμε να έχουμε αυτοκίνητα και πιο οικολογικές μεταφορές με κανόνες, με ωράρια τα οποία ε, ουσιαστικά θα είναι και σημεμένα, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση για να έχουν ευελιξία αυτές οι περιοχές. Μπορούμε να δώσουμε λοιπόν ένα πολύ πιο κοινοτόμο χαρακτήρα σε αυτές τις αεροκατοικημένες περιοχές. Μπορούμε να βρούμε ε, ουσιαστικά μεγαλύτερη συμμετρία, να μην υπάρχουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις όπως είδαμε στην τελευταία παρέμβαση. Και εγώ Πιστεύω ότι μια επικράτεια που δεν έχει κινητικότητα είναι πιο φτωχή, πιο αποκλεισμένη και σε αυτές ε, τις ε, περιοχές όπου ζουν ηλικιωμένοι άνθρωποι, άνθρωποι με αναπηρίες, γυναίκες, άνθρωποι ε, με οικονομικές δυσκολίες που δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Εδώ λοιπόν πρέπει να βρούμε τη λύση, να σχεδιάσουμε τις αστικές πολιτικές και πριν να δώσουμε τα κονδύλια να ξέρουμε ακριβώς πώς και πού θα δαπανίσουμε και με ποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να προωθήσουμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τέλες, κυρία Λαντέν, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σουηδικά. Καταρχάς θα ήθελα να συμφωνήσω ότι πρέπει να εξετάσουμε το σύστημα μεταφορών στο σύνολό του και να εξετάσουμε όλα τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό, είτε είναι ποδήλατα, μεγάλα λεωφορεία ή οι δημόσιες μεταφορές κατόπιν ζήτησης, όπως σας ανέφερα πριν. Αυτό ισχύει και ε, στις ε, μεγάλες πόλεις όπου έχουμε μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού και ευκαιριών. Ε, είναι δύσκολο να δούμε πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε την τάση αυτή. Πώς μπορούμε να δώσουμε σε όσο γίνεται περισσότερους πολίτες να ε, εκμεταλλευτούν ε, αυτές τις προσφορές που δίνονται χωρίς ε, να πρέπει να μετακινούνται κάθε μέρα στα μεγάλα αυτά κέντρα. Αρκετοί μίλησαν και για την ανάγκη υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εφαρμοστούν ε, τέτοιου είδους ε, λύσεις. Ε, το πρώτο που μου έρχεται εμένα στο νου είναι η ανάγκη υποστήριξης για τα πιλωτικά προγράμματα για να δοθούν διάφοροι τρόποι και στο Βέρμπλαντ και σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ώστε να μπορούν να δοκιμαστούν ε, λύσεις που δεν ξέρουμε αν τελικά θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δυστυχώς ε, είναι πολύ περιορισμένοι οι πόροι τη σημερών ημέρα. Και έτσι φτάνω και στην άλλη έκκληση, της ευέλικτες λύσεις Πολύ σημαντικό είναι το θέμα της εμπιστοσύνης των πολιτών ότι θα λειτουργήσει τελικά το σύστημα αυτό και να κατανοήσουν καλά το σύστημα. Ε, μπορεί να χρειαστούν ε, ε διάφορα προγράμματα κατάρτισης ε, και μπορεί να φαίνονται πολύ εύκολες οι λύσεις ε, με εφαρμογή στο κινητό. Ε, αυτό ισχύει για τους περισσότερους, όχι όμως για όλους. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει εναλλακτική λύση για τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους βοηθήματα. Κυρία Πρόεδρε, και εσείς θέσατε την ερώτηση σχετικά με το πώς βλέπουμε τις ε, δωρεάν ε, μεταφορές. Ε, είναι πολιτικό το θέμα αυτό. Υπάρχουν ωστόσο κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να τονίσουμε. Υπάρχει ένα πολύ πρακτικό θέμα. Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι υποδομές, το εισόδημα από τις μεταφορές στο Βέρμλαντ είναι περίπου ε, οι δαπάνες μάλλον στο Βέρμλαντ είναι 200 εκατομμύρια ε, το χρόνο. Για το σύνολο της Σουηδίας είναι 40 δις ε, κορώνες και δεν καλύπτονται και όλες οι δαπάνες αυτές από τα εισιτήρια. Είναι λοιπόν πολιτικό το θέμα. Επίσης υπάρχει και μια άλλη πτυχή. πολύ συχνά ε, γίνονται λιγότερο ελκυστικές ε, οι μαζικές μεταφορές και προτιμάει τελικά ο κόσμος να πάρει το αυτοκίνητο. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε καλές μαζικές μεταφορές ως πραγματική εναλλακτική λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λάντιν. Κύριε Στέρμπα, τώρα έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω σημειώσει εδώ πέρα κάποιες ε, ερωτήσεις. Ε, ένα πρόβλημα είναι, ε, αν το πρόβλημα είναι ότι μας λείπουν οι καινοτομίες ή αν μας λείπει η χρηματοδότηση. Στην κεντρική βοημία το πρόβλημα των ε, καινοτομιών μπορεί να λυθεί εύκολα και να χρηματοδοτηθούν, για παράδειγμα με ευφυή e συστήματα ε, εισιτηρίων. Είναι ένα σύστημα πώλησης ε, εισιτηρίων. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί, να υλοποιηθεί και έχουμε σημειώσει πρόοδους όσον αφορά την ψηφιοποίηση. Από την άλλη υπάρχουν συστήματα όπως είναι τα νέα, ε, τα νέα συστήματα πρόθεσης των αυτοκινήτων ε, με μπαταρίες για παράδειγμα. Ε, υπάρχουν όμως ε, κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά την χρηματοδότηση. Το πρόβλημα είναι να μην περιορίζεται τόσο η κυκλοφορία ώστε να υπάρχουν απώλειες στον προϋπολογισμό των επιχειρήσεων. Είναι σημαντικό να υπάρχει επαρκής ε, χρηματοδότηση για τακτική ανανέωση του στόλου. Θα πρέπει οι δημόσιες ε, μεταφορές να είναι ελκυστικές για τους περισσότερους πολίτες και όσον αφορά τα νέα συστήματα προώθησης θα πρέπει να συμβάλλουν ε, στον οικολογικό προσανατολισμό των ε, μεταφορών ε, ε, στους περιοχές όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σιδηρόδρομος. Άλλο θέμα είναι η χρήση οχημάτων σαν τραμ. Τρόλεϊ για παράδειγμα ή τραμ ε, εδώ είναι το θέμα της ε, ηλεκτροδότησης. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις αστικές αρχές, ε, τις σιδηροδρομικές και την τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως είπα στην παρουσίασή μου, θα πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό και δεσμευτικό σχέδιο Στην ε, Τσεχία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 13 ε, περιφέρειες και η πρωτεύουσα της Πράγας. Ε, κάθε περιφέρεια έχει δικό της σχέδιο μεταφορών και πέρα από την πρωτεύουσα υπάρχει διαφορετικό σύστημα εισιτηρίων και δεν είναι συμβατά μεταξύ τους. για να το πω χοντρά, εάν ε, θέλει κάποιος ε, να ταξιδέψει σε όλη την Τσεχία, που είναι και σχετικά μικρή χώρα, θα χρειαστεί 10 διαφορετικά εισιτήρια. Και αυτό σίγουρα αποτελεί αντικίνητρο. Θα πρέπει να εξετάσει ο επιβάτης σε τι εισιτήριο πρέπει να πληρώσω, τι ε, προϋποθέσεις ισχύουν για το κάθε είδος μεταφοράς. Ανάμεσα λοιπόν στις διάφορες περιφέρειες υπάρχουν προβλήματα. Άλλο θέμα είναι το πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε σιδηρόδρομους ε, που να ξεπερνάνε τα όρια των διαφόρων περιφερειών. Κανείς δεν θέλει να χρηματοδοτήσει κάτι το οποίο θα ε, χρησιμοποιηθεί σε άλλη περιφέρεια. το κράτος ε, θα πρέπει να υπαγορεύσει να υπάρχουν ε, συνδέσεις ανάμεσα στις διάφορες ε, περιφέρειες. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει απλοποίηση όσον αφορά τα εισιτήρια και αυτό δυστυχώς αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τους ταξιδιώτες και όσον αφορά την μαζική μετανάστευση προς κάποιες περιοχές. Βλέπουμε συγκέντρωση του πληθυσμού στην Πράγα και σε άλλα μεγάλα κέντρα, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις και χωρίς να έχει δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή. Σήμερα, όταν πηγαίνει κανείς στη δουλειά του, βλέπει ουρές αυτοκινήτων κάθε μέρα και μάλιστα όλη τη μέρα. Δεν είναι καν κάτι που ισχύει μόνο κάποιες ώρες αιχμής το πρωί και το απόγευμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει επηρεάσει θετικά τη σύγκληση των νέων κρατών μελών διότι συγχρηματοδοτεί ε, πολυτροπικούς ε, διασυνοριακούς διαδρόμους. Βλέπουμε πολύ καλή πρόσβαση προς τις, ε, περιφέρει... προς τις πρωτεύουσες, αλλά ε, οι περιοχές που απέχουν από αυτές τους διαδρόμους είναι απομονωμένες. Ε, στην καλύτερη περίπτωση εξαρτώνται οι άνθρωποι εκεί από λεωφορεία ή στη χειρότερη περίπτωση από δικό τους ιδιωτικό αυτοκίνητο. Και βλέπουμε απαρχαιωμένα αυτοκίνητα και άλλα προβλήματα. Και πέρα από τα ε, διευρωπαϊκά δίκτυα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί στις ε, περιφερειακές υποδομές και τις ε, ε, διαπεριφερειακές συνδέσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν ποιοτικά δίκτυα σιδηροδρόμων και θα πρέπει να ιεραρχήσουμε σωστά τις υποδομές όσον αφορά τις μεταφορές μεταξύ των περιφερειών, ε, τις ε, τοπικές μεταφορές, όλα αυτά θα πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους. Ε, και υπάρχουν εμπειρίες από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, όπου υπάρχει τρένο υψηλής ταχύτητας. Εμείς θέλουμε οι αυτοκινητόδρομοι να μην ε, συνδέουν μόνο ε, μεγάλες πόλεις, ε, αλλά και διάφορες περιφέρειες. Οι περιφέρειες να μπορούν έτσι να βρεθούν πιο κοντά εντό αγωγικών στις περιοχές συγκέντρωσης του πληθυσμού. Εάν συμβεί αυτό, δεν θα χρειάζεται οι άνθρωποι να μετακομίσουν στις μεγάλες πόλεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ας ακούσουμε τώρα τον τελευταίο μιλητή, τον κύριο Κρίστιανς, για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ και πάλι, κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μια μαγική ενία λύση για όλους. Είναι πολύ σχηδές, πολύπλοκο το πρόβλημα και θα πρέπει από κοινού να συνεργαστούμε σε διάφορους τομείς πολιτικής για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ενδεχομένως όμως και μάλλον αυτό είναι περισσότερο, αν θέλετε, επιστημονική έννοια, έχει αποτελέσει και αντικείμενο πολυπιλωτικού προγράμματος, ανάπτυξη οικονομική που να έχει ως βασικό γνώμονα τις μεταφορές. Η έννοια αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει και στην πράξη, γιατί ουσιαστικά είναι κάπως αυτοματοποιημένη, έχει μια αυτοματοποιημένη συνιστόσα αποκεντρικοποίησης. Ουσιαστικά να πτήσει κανείς υπηρεσίες στέγασης και διάφορες άλλες υπηρεσίες βάση του δικτύου μεταφορών. Κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργίες και υπηρεσίες αυτόματα δημιουργούνται, αλλά χρειάζεται και μια κριτική κρίσιμη μάζα. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη σε ένα χωριό. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι όταν δημιουργήθηκαν τέτοια πιλωτικά προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης βάσει των μεταφορών, είχαμε και φαινόμενα αύξησης των τιμών, όπως για παράδειγμα συστέγαση, στέγαση, συγκέντρωση ενός πιο ευκατάστατου πληθυσμού. Τώρα, θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε διαφορετικές πολιτικές, για παράδειγμα υπηρεσίες στέγασης γύρω από συγκεκριμένες περιοχές, γύρω από, συγκεκριμένες, από συγκεκριμένα χωριά ή αεροκατοικημένες περιοχές και ενδεχομένως να έχουμε έτσι και καλύτερα δίκτυα μεταφορών. Τώρα όσον αφορά τι ελεύθερε δημόσιε κοινωνίε. Απλή η έννοια αυτή και μ' αρέσει, αλλά δυστυχώ οτιδήποτε είναι δωρεάν οδηγεί σε υπερκατανάλωση και δεν πρέπει να έχουμε εμεί τώρα κάτι τέτοιο εδώ. Χρειαζόμαστε μια κατανάλωση μεταφορών η οποία να είναι καλή και βιώσιμη, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το σύστημα αυτό των ελεύθερων δημόσιων συγκοινωνιών ω προσωρινή τουλάχιστον λύση. Για να απαντήσω και στον κύριο Ντάνιελσον, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε θεωρώ αν χρειαζόμαστε μάλλον ε, χρηματοδότηση ή άλλες λύσεις, ευέλικτες λύσεις ήδη υπάρχουν. Αλλά η αγορά εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουμε. Αν δείτε πώς έχουν τα πράγματα στις Βρυξέλλες, είναι πολύ πιο διαφορετικά τώρα από ό,τι ήταν πριν δύο χρόνια. Έχουμε ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα, ηλεκτροκίνητα, ποδήλατα. Η αγορά έχει ήδη εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από δειτε πώ εμείς στι βρυξελλες ίδιοι. Οι λύσεις θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν. Η Ευρωπαϊκή οτι εμεί οι ιδιοι οι λύσει θεωρω μπορεί να δραματίσει ένα καθοριστικό ρόλο ρυθμίζοντα το οικονομικά προσιτό, την προσβασιμότητα των ε, μέσων αυτών μεταφοράς. Οι νέες αυτές αναδυόμενες ε, λύσεις ε, πολλές φορές επισπεύδουν πολύ συχνά και τα προβλήματα. Για παράδειγμα, στις Βρυξέλλες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο τα ηλεκτρονικά πατίνια. Ποιος τα χρησιμοποιεί όμως, ε, κυρίως άνθρωποι με χαμηλό εισόδημα και ξέρετε ότι ήδη ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ έντονος στον τομέα αυτό. Εμείς μπορούμε να ρυθμίσουμε κάπως τη χρησιμοποίηση των νέων αυτών καινοτόμων μέσων μεταφοράς. Τώρα, τα ποδήλατα και τα ηλεκτρονικά ποδήλατα, 25 χιλιόμετρα μπορεί να τα κάνει κανείς πολύ εύκολα με ένα ηλεκτροκίνητο ποδήλατο, ακόμα και δεν έχει κανείς μια άριστη σωματική κατάσταση. Στη δική μου σχολεία ε, εκπαίδευσης ε, στην ποδηλασία βλέπουμε ότι τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα αποτελούν πραγματικά λύση για πάρα πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας. Κάποια σχέδια κυκλικής οικονομίας, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τράπεζες για παράδειγμα που μπορούν να μισθώσουν κάποια ηλεκτροκίνητα ποδήλατα. Τα ποδήλατα αυτά μετά από ένα χι χρονικό διάστημα μπορούν να έλθουν σε εμά και να τα χρησιμοποιήσουμε εμεί στο δικό μα το επίπεδο. Νομίζω ότι τέτοια παραδείγματα μπορούμε να ακολουθήσουμε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση πάντα αποτελεί πρόβλημα για όλου. Χρειαζόμαστε ένα αρχικό κεφάλαιο για να ξεκινήσουν διάφορε ιδέε, αυτό ισχύει, αλλά α αφήσουμε έπειτα και την αγορά και τους κοινωνικού επιχειρηματίες να λάβουν δράση, Α τους δείξουμε πού χρειάζονται επενδύσεις, πού πρέπει να επενδύσουν και α τους αφήσουμε να επιλέξουν ελεύθερα. Για μία ακόμη φορά θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε τα βιώσιμα αυτά σχέδια αστική κινητικότητα. Πάρα πολλά πράγματα έχουν ήδη γίνει σε επίπεδο πόλεων, αλλά αυτή η συμμετοχική προσέγγιση, η επιμερισμένη κινητικότητα ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί στις ομάδε χαμηλού εισοδήματο. Δεν έχουμε στοχεύσει καλά τι ομάδε αυτέ, ούτε εκπροσωπούνται αρκετά ακόμα σε αυτά τα project που έχουν να κάνουν με την αστική κινητικότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλες σας τις παρεμβάσεις. Απλώς να πω πως όταν μιλάμε για δωρεάν μεταφορές, δεν είναι δωρεάν, είναι η χρήση που γίνεται, που είναι δωρεάν, γιατί κάποιος πληρώνει όπως και να έχει για τις μεταφορές και ποιος πληρώνει οι πολίτες με τους φόρους τους. Έτσι λοιπόν όταν ε, λέμε κυρία Ντάλη, δωρεάν μεταφορέ τίποτα δεν είναι δωρεάν, η χρήση είναι δωρεάν. Σας ευχαριστώ για την εμπειρογνωμοσύνη σας και που μας παρουσιάσατε τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε και ταυτόχρονα το είπατε, πρέπει και εμέσως να κινηθούμε για να προωθήσουμε την κινητικότητα στην Ήπεθρο. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία, αλλά θα πρέπει και ο κάθε ε, φορέας, ε, ο κάθε ερμόδιος να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία, να τα κάνει δικά του. Δεν υπάρχουν μαγικά εργαλεία, παρόλα αυτά θα πρέπει να γίνουν προσβάσιμα σε όλους. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας, να χειροκροτήσουμε τους ομιλητές μας. Και δυστυχώς ε, θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Εγώ θα σας ε, πω εις το επανειδήν και όσοι ενδιαφέρονται για τις διαφάνειες μπορούμε να σας τις στείλουμε. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να διακόψω εδώ τη συνεδρίαση γιατί θα τα ξαναπούμε στις 5 για τη συνεδρίαση των συντονιστών. Συμφωνείτε κύριε Ντάνιελσον. Φαίνεστε ενθουσιώδης. D'accord, très bien. La séance est levée. Διακόπτεται η συνεδρίαση. Θα τα ξαναπούμε στις 5 στην ίδια αίθουσα.